el señor presidente. Άρχεται η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση του κυρίου Κάμπρνοχ για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και για τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο εισηγητής